της έκθεσή μου και ευελπιστώ ότι στην αυριανή ψηφοφορία θα καταφέρουμε να εγκρίνουμε την έκθεσή μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σιγητά. Θα ήθελα και εγώ να σας ε, επενέσω για, το, για την έκθεση και να πω ότι όταν ήμουν μέλος ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, συζητούσαμε για τη βία σε αθλητικές εκδηλώσεις ε, στα ποδοσφαιρικά γήπεδα και μερικές εκθέσεις ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης για το θέμα αυτό θα μπορούσαν να γίνουν αντικείμενο μελέτης ε, και να τροφοδοτήσουν τη δική μας συζήτηση. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Ολοκληρώνουμε τη συζήτηση για την έκθεση του κυρίου Φίσας και περνάμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσης διάταξης της παρεμβάσης ενός λεπτού. Ο κύριος Κούκαν, πρώτος για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε κοινέ αξίε, δικαιώματα και υποχρεώσει. Αυτή ήταν η ιδέα πίσω από την ίδρυση τη Ένωση και μόνο με την ιδέα αυτή μπορεί να λειτουργήσει και να εξακολουθήσει να λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θεωρούμε ότι η Ουγγαρία αποτελεί σημαντικό εταίρο. Ο εταίρο αυτό έχει αποδείξει ότι αποτελεί και αναπόσπαστο μέλο τη Ευρωπαϊκή οικογένεια. Είναι λοιπόν απαραίτητο να το ξεκαθαρίσουμε πραγματικά αυτό. Στην παρούσα χρονική φάση διεξάγεται μια συζήτηση με την Ουγγαρία για την ανεξαρτησία της Εθνικής Τράπεζας και του δικαστικού σώματος και για θέματα τα οποία είναι κατοχυρωμένα στις ευρωπαϊκές συνθήκες, όπως για παράδειγμα τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν πρέπει να υποτιμούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτά. Είμαι βέβαιη ότι όλοι επιθυμούμε η Ουγγαρία να είναι ισχυρός εταίρο ο οποίος θα σέβεται τις κοινέ αξίες και ελπίζω αυτό να επιθυμεί και η, Ευρωπαϊκή, και η Ουγγαρία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε πρόεδρο Και ο επόμενος ομιλητής είναι, είναι ο κύριος Ιβαν. Για ένα λεπτό. Παν Για ένα λεπτό έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας ε, στο γεγονός ότι ε, ασχοληθήκαμε αυτές τις μέρες με δύο πολύ σημαντικές συνθήκες που θα επηρεάσουν τη ζωές μας με πολύ ριζικό τρόπο. Θα επηρεάσουν και την καθημερινότητα και την ιδιωτική ζωή των ε, πολιτών αλλά και το επίπεδο απασχόλησης και το βιωτικό επίπεδο σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εξετάστηκαν καν αυτές οι συνθήκες, η ΆΚΤΑ και οι άλλοι. Και, ορισμένες, και ορισμένοι αρχηγοί κρατών δεν έθεσαν καν ε, το ζήτημα αυτό στις εθνικές βουλές. Ε, δεν γνωρίζει κανείς στη Ρουμανία τι σημαίνει άκτα ή τι σημαίνει σύμφωνο σταθερότητα. Αυτό είναι δημοκρατία. Όχι. Αν θέλουμε να θέσουμε ένα τέρμα στην κρίση και θέλουμε μια ενιαία, ενωμένη και ισχυρή Ευρώπη, θα πρέπει να εφαρμόσουμε και μπράκτο στι δημοκρατικές αξίες κυρία Μπιλμπάου. Ευχαριστώ. Μεταξύ της δεκαετίας 60 και 80 απήχθησε στην Ισπανία χιλιάδες παιδιά και οι μητέρες ενημερώθηκαν ψευδώς ότι τα παιδιά τους είχαν πεθάνει και μάλιστα πιστοποιήθηκαν θάνατοι ενώ στην ουσία απήχθησαν και ε, πουλήθηκαν αυτά τα παιδιά. 600 τέτοια παραδείγματα, κρούσματα είχαμε στη χώρα των Βάσκων. Έχουν ανοιχτεί μέχρι στιγμή τρει τάφοι, ήταν ε, κενή και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιος μπορούσε να ε, διαπράξει αυτά τα αυτά τα εγκλήματα. Μέχρι στιγμής ίσχυε σιωπή. Τώρα αρχίζουν οι οικογένειες να ψάχνουν τα παιδιά τους και να ζητούν αποκατάσταση και δικαιοσύνη. Είχαμε χιλιάδες ε, προσωπικές τραγωδίες που δεν μπορούν να αποκατασταθούν. Είναι ανεπανόρθωτες αυτές οι ζημιές και οι βλάβες και οι ψυχικές ε, που επηρεάζουν και τις φυσικές οικογένειες και τις βιολογικές, τις βιολογικές οικογένειες και τις οικογένειες που έχουν υιοθετήσει αυτά τα παιδιά. Θα πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια για να διαλευκανθούν όλες αυτές οι υποθέσεις. Ο κύριος Τρεμόπουλος. Απουσιάζει ο κύριος Ταβάρες. Απουσιάζει ο κύριος Φερέιρα. Ευχαριστώ. Τα στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύθηκαν για την ε, ανεργία ουσιαστικά απαγγέλουν κατακορητήριο κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ε, Πορτογαλία έχουμε ανεργία 14%, 31% ανεργία των νέων. Ε, άνευ τα στα 30 χρόνια της δημοκρατίας. Είναι δραματικές οι ε, συνέπειες της εφαρμογής ε, του προγράμματος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανεργία, ε, πλήττουμε τις ε, στρατηγικές ε, πτυχές της οικονομίας, την υγεία, την κοινωνία. Έχουμε όλο και μεγαλύτερη φτώχεια. Και η καινή ρητορική της ανάπτυξης και της απασχόλησης ε, πέφτουν στο κενό. Ενώ ταυτόχρονα το εξωτερικό χρέος και το άλοθη που χρησιμοποιούμε για το πρόγραμμα λιτότητες ε, θα συνεχιστούν το 2012 και θα οδηγήσουν σε ακόμη μεγαλύτερη ενεργεια και σε ακόμη μεγαλύτερο χρέος. Αυτό είναι, αυτός είναι ο δρόμος που οδηγεί αναπόφευκτα στον όλεθρο. Ο όλεθρος που μπορεί να αποφευθεί με διαφορετικές πολιτικές. Αυτό ζητούν ε, οι συμπολίτε μα και στην Πορτογαλία και σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλαγή τη πολιτική. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριο Ζόμπρο. Κύριε Πρόεδρε. Ε, το Νοέμβριο είχα υποβάλει μια ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 18 Νοεμβρίου για το ΑΚΤΑ ε, για ένα πολύ σημαντικό θέμα που είναι συγκινησιακά φορτισμένο στη δημόσια συζήτηση σε πολλές χώρες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Πολωνία. Ρώτησα μεταξύ άλλων και το εξής την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το άκτα ε, τηρεί τις θεμελιώδεις δεσμεύσεις και τις νομικές διατάξεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 5 Ιανουαρίου έλαβα απάντηση από τον Επίτροπο Καλ Ντεγκούχτ εκ μέρου ευρωπαϊκή Επιτροπή και μου είπε ναι, το, η άκτα ε, συνάδει με την ε, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, είναι νομότυπη με τις ε, νομικές διατάξεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, στις 24 Νοεμβρίου είχαμε την νομολογία του ΔΕΚ που προβλέπει ότι η άκτα δεν είναι καθόλου νομότυπη. Ορισμένα στοιχεία της άκτα παραβιάζουν θεμελιώδη δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια διαλεύκαση του κατά πόσο η άκτα είναι όντω νομότυπη και συνάδει με το κοινωτικό δίκαιο και τι θεμελιώδει ελευθερίε. Ο κύριο Χάρτονγκ έχει το λόγο. Δεν τον βλέπω, ο κύριο Μπίνα. not, and Ούτε αυτό είναι εδώ, ο κύριο Σικέρσκι. Το 2011 ήταν μια χρονιά με πολύ σημαντικά γεγονότα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε το, το Fiscal Pact, το Δημοσιονομικό ε, Σύμφωνο, πολύ σημαντικό. Επίσης, ε, συζητήσεις για, τις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 2013-2020. Είχαμε και την πεντηκονταετία της κοινή γεωργικής πολιτικής, μια πολύ σημαντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε και πολύ σημαντικές προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε ε, το χρόνο αυτό. Ε, είχαμε την αύξηση των αγαθών ε, των πρώτων υλών και μείωση ταυτόχρονα του γεωργικού εισοδήματος. Υπάρχουν πολλά προβλήματα γιατί εκτοξεύθηκαν οι τιμές τροφίμων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πολύχρονη εμπειρία μας από την ΚΑΠ ήταν πολύ πλούσια και χρειαζόμαστε σίγουρα ενημερωτικέ εκστρατείες στα πλαίσια της αναθεώρησης γιατί νομίζω ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε την γεωρική πολιτική και τη συνέχισή της και για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, μέχρι το 2020 δηλαδή. Σας ευχαριστώ. Το λόγο κυρία Φλασίκοβα. Δεν είναι εδώ. Ο κύριος Κορτές. Ευχαριστώ. Η πολυεθνική ΤΕΚΑ μίλησε για απολύσει 198 υπαλλήλων στο Κάχο, Σαταντέρα και Κατάβρια. Είναι σημαντικό το πρόβλημα της ενεργείας. Επίσης, άλλες 400 θέσεις απασχόληση θα χαθούν από θηγατρικές της ΤΕΚΑ. Η ΤΕΚΑ δεν έχει επαρκείς και αποχρόντες οικονομικούς λόγους για τις απολύσεις αυτές. Απλώς θέλει να μετακατασταθεί εκτός Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει από την Κατάβρια και την Ισπανία μεγαλύτερη προστασία των εργαζομένων, ε, βρίσκοντας οριστική λύση σε αυτή σε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα και να διερευνηθούν όλες οι δυνατότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ίσως και ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου ε, Παγκοσμιοποίησης. Δεν, έχουμε, δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλους ανέργους. Άλλωστε η τοπική διοίκηση της Καντάβρια είχε ε, προεκλογικά ε, υποσχεθεί να εγγυηθεί τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ας το κάνει, γιατί πραγματικά αυτή είναι το, ο βιομηχανικός ιστός της περιοχής Καντάβριας. Θα πρέπει οι εργαζόμενοι να τύχουν προστασίας. Ευχαριστώ κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην Αρλινδία λέμε ότι αν είμαστε πειθαρχικοί στα δημοσιονομικά θα αποφύγουμε μελλοντικέ κρίσεις. Από το 2002 μέχρι το 2008 η Ιρλανδία δεν έσπασε ποτέ το πακέτο σταθερότητας αντίθετα με άλλες χώρες. Ξέρουμε λοιπόν ότι ο σεβασμός των κανόνων δεν είναι πάντα αυτό το οποίο χρειάζεται ιδιαίτερα σε σχέση με την παρούσα χρήση. Είχαμε μια σχέση ΑΕΠ και χρέους 20%. Το 2014 θα έχει πάει στο 145%. Καμία αναπτυγμένη οικονομία δεν μπορεί να αντέξει τέτοιου είδους χρέη. Εμείς ζήσαμε τέσσερα χρόνια λιτότητας. Εμείς έχουμε υψηλό χρέος γιατί εξαγοράσαμε τα χρέη των τραπεζών αλλά παρόλα αυτά μας λένε ότι τα ίδια θα γίνουν χωρίς ευρωομόλογα, χωρίς άλλα προγράμματα σωτηρίας της οικονομίας μας. Νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με ένα κάποιο εκβιασμό εδώ σε σχέση και με την επικύρωση της συνθήκης εφόσον θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει την πολιτική της, την οικονομική και για τον ίδιο της τον εαυτό και για τη δική μου χώρα. Ευχαριστώ. Μετά την επιβολή στην Ελλάδα από το Βερολίνο ενός τεχνοκράτη ως πρωθυπουργού, η δήλωση η Γερμανία ότι η χώρα χρειάζεται και Υπουργό Οικονομικών που δεν θα είναι Έλληνα. Δεν ξέρει η κυρία Μέρκελ ότι το χειρότερο μπορεί να κάνει κανεί ένα λαό είναι να τον ταπεινώνει και να τον υποχρεώνει να, δέχεται, να γίνεται υποτελή. Στην εποχή Μπρέσνευ στη Σοβιετική Ένωση ε, αναφερόταν ε, το αστείο ότι το τρένο της ε, Επανάστασης έχασε την ατμομηχανή του και ζητούσε από τους επιβάτες να πηδήξουν. Τελικά αυτό συμβαίνει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας λένε ότι θα πρέπει να εφαρμόζουμε μονίμως την ίδια συνταγή παρά την αποτυχία που έχει δείξει στην εφαρμογή της. Θα πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξουν τα πράγματα και ακόμη και στις αγορές μια μέρα να σταματήσουμε επιτέλους να προσποιούμαστε. Ο κύριος Παπα-Νικολάου, επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν χρειάζεται να υπενθυμίσω πόσο κρίσιμες είναι οι επόμενες ημέρες, αν όχι οι επόμενες ώρες, για την οριστική αντιμετώπιση της ελληνικής κρίσης χρέους Χρειάζεται όμως να υπενθυμίσω ότι στις δύσκολες αυτές στιγμές όλοι πρέπει να κάνουν ό,τι είναι δυνατό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Αυτό κατά τη γνώμη μου πρέπει να κάνει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Να κάνει δηλαδή την κίνηση που θα ανακούφιζε κατά 10 τουλάχιστον δισεκατομμύρια ευρώ το δημόσιο χρέος της Ελλάδος, δεχόμενη το ανάλογο κούρεμα στα ομόλογα που κατέχει. Και προσοχή, δεν ζητάω από τον κύριο ντράγκη να υποστεί ζημιές η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα ζητάω απλώς να μην προσποριστεί κέρδος γιατί όταν η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα αγόρασε τα ελληνικά ομόλογα στο 75% της αξίας τους περίπου στη δευτερογενή αγορά και αναμένει στη λήξη τους να πληρωθεί στο 100% τι άλλο παρά κέρδος μπορεί να χαρακτηριστεί αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο επόμενο η κυρία Γιάλα Σέντερ. Ε, χρεοκόπησε από τη μια στιγμή στην άλλη αφήνοντας ε, απεγνωσμένους 2.000 ε, εργαζόμενους και 20.000 επιβάτες χωρίς καμία αποζημίωση και χωρίς καμία ενημέρωση. Όλοι αυτά τα θύματα κακής διαχείρισης εργοδοτών που είχαν συνηθίσει να είναι κρατικοδίαιτοι και να μην διαχειρίζονται καλά τα κρατικά κονδύλια. Επίσης είχαμε επιδοτήσεις αναπατελεσματικές Κατηγορήθηκε μερικές φορές ακόμη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμεί λέμε όμως ότι ήδη το 2009 είχαμε ζητήσει νομοθετικά μέτρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αυληθούν οι συνέπειε χρεοκοπία αεροπορικών εταιριών και να προστατευτούν οι εργαζόμενοι τους, οι επιβάτες και να εφαρμοστούν και κάποιες διαδικασίε για την προστασία των εργαζομένων σε τέτοιε περιστάσει. Ζητούμε, κύριε Επίτροπε, μια νομοθετική πρόταση, όχι μόνο προαιρετικές ε, διαδικασίες. Θα πρέπει να προστατεύσουμε και τους εργαζόμενους και τους ε, επιβάτες που δεν αξίζουν πραγματικά τέτοιες τύχη και μεταχείρισης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπουσόη. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Τον Ιανουάριο πολύ. Ε, Ρουμάνοι βγήκαν στους δρόμους και έχουν μείνει στους δρόμους έκτοτε. Δεν μπορούμε να διαφορήσουμε στις φωνές τους. Γιατί οι πολίτες αυτοί θέλουν να ζήσουν σε μια χώρα όπου οι εκλογές δεν διοργανώνονται μόνο προς όφελος του κυβερνητικού κόμματος. Ο κόσμος αυτός ε, που ζει σε μια ευρωπαϊκή χώρα όπου δεν περνάνε οι νόμοι Περνώντα από το Κοινοβούλιο, με την έγκριση του Κοινοβουλίου και ο κόσμο αυτό θέλει ένα σύστημα που δεν αλλάζει, για παράδειγμα, το υγειονομικό σύστημα σε μία νύχτα, όπου δεν ε, λαμβάνει αύξηση μισθού για να δει αύξηση και των ε, τιμών μετά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας τις συνέπειες της πολιτικής λιτότητας και περιορισμού των κρατικών δαπανών στην Ισπανία και η κεντρική κυβέρνηση και με η τοπική αυτοδιοίκηση συρρυκνώνουν δραστικά τις δημόσιες δαπάνες, στην υγεία, την εκπαίδευση, κάτι που επιδεινώνει και την δημόσια υγεία και το σύστημα της εκπαίδευσης και δίνει λαβές για ιδιωτικοποίηση της υγείας και της εκπαίδευσης. Αυτό είναι απαράδεκτο σε, μια, σε ένα μικρό δήμο της Καταλωνίας αυτή τη στιγμή ε, προσπαθούν να κλείσουν ε, το κέντρο παροχής ε, πρώτων βοηθειών και μάλιστα οι εργαζόμενοι ήδη 97 μέρες έχουν κάνει κατάληψη για να αποφευθεί το κλείσιμο αυτού του κέντρου οι πολίτες έχουν κινητοποιηθεί, έχουν κινητοποιηθεί για να προσθέσουν κάτι που είναι δικό τους. Ε, θέλουν κοινοφελείς ε, ποιοτικέ υπηρεσίες στην υγεία και στην εκπαίδευση. Σας ευχαριστώ. presa κύριος Νικολέσκου. Ευχαριστώ μου. Έκανε εντύπωση βλέποντας τις ε, εφημερίδες της πρωινές ένα ξενοφοβικό ε, καρτούν το οποίο προετοίμασε ή σε ένας υποψήφιος του Εθνικού μετόπου Βρίζει ασύστολα τους Ρωμάνους, χρησιμοποιεί λέξεις που δεν θέλω να χρησιμοποιήσω. Είπε ε, πρέπει να φοβάστε ακόμα και τους Ρωμάνους Αγιοβασίλιδες, οι οποίοι θα σας κλέψουν ακόμα και την τηλεόραση. Ε, ε, είναι απαράδεκτο να βλέπουμε τέτοια πράγματα, ιδιαίτερα για μια χώρα η οποία πάντα στήριζε τη Γαλλία και τις γαλλικές αξίες. Περιμένουμε από τους ηγέτες του Εθνικού Μετώπου να καταδικάσουν τη συγκεκριμένη αυτή γελιογραφία. Κυρία Κρέτου. Πρόεδρε, η κατάσταση πολιτική στη Ρουμανία είναι πολύ ε, περίπλοκη και οι βασικές αρχές του κράτους δικαίου αγνοούνται. Τα τελευταία χρόνια τα πράγματα χειροτερεύουν, ο κόσμος διαδηλώνει, διαμαρτύρεται, η παρούσα κυβέρνηση είναι πραγματικά απαράδεκτη, έχει δημιουργήσει πάρα πολλά κοινωνικά προβλήματα, έχει αγνοήσει συστηματικά το κοινοβούλιο, έχει απαγορεύσει τον πολιτικό πλουραλισμό έχει εφεύρει ψευδή πολιτικά κόμματα νέα για να τη στηρίξουν. Συνεπώς η αντιπολίτευση αποφάσισε να αρνηθεί να συνεχίσει να λαμβάνει μέρος της εργασίες της Ρωμανικής Βουλής γιατί τα δικαιώματα της αντιπολίτευσης πλέον δεν διασφαλίζονται. Next speaker is Mrs. Mr. President, the European Parliament came under a cyber attack. Η κυρία ευχαριστώ Πρόεδρο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέστη μια κυβερνοεπίθεση την προηγούμενη εβδομάδα μετά από την υπογραφή μια σχετική συμφωνία με την Ιαπωνία. Εν τω μεταξύ έλαβα μεγάλο τμήμα μηνυμάτων από Ευρωπαίου πολίτε που ανησυχούν για τα δικαιώματά του και θεωρώ ότι είναι περίεργο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 22 από τα κρατημέλη τη υπέγραψαν την άκτα πριν να αντιμετωπίσουν τι ανησυχίε των πολιτών με κατάλληλο, διαφάνη τρόπο, όπω πρέπει να γίνεται σε δημοκρατίε. Γι' αυτό, λοιπόν, καλά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να αυξήσουν τι προσπάθειε για να ενημερώσουν του πολίτε για το άκτα, για να υπάρχει και στην κατάθεσή του όταν επικυρωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το άκτα δεν θα ε, παραβιάσει τα βασικά δικαιώματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα για την ελευθερία έκφραση. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο, ο κύριο Σόγκορ. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά το νέο Ουγγρικό Σύνταγμα, ακούστηκε ε, φωνές κριτικής από πολλές πλευράς προς την ε, Ουγγρική κυβέρνηση. Δεν θα ήθελα να επισέλθω σε σημεία τέτοια της ε, κριτικής. Ως εκπρόσωπος της Ουγγρικής μειονότητας στην Ρουμανία. Παρακολουθώ και θέματα ιστορικής πολιτικής της Ρουμανίας, Ουγγαρίας, Σλοβακίας και Σερβίας. Συνάδελφοι, αν ε, ανησυχείτε για τα δικαιώματα των μειονοτήτων, να σας ε, επιστήσω ότι γίνεται την προσοχή σχετικά με το τι γίνεται με τις επίσημες γλώσσες στην Σλοβακία και σε ό,τι αφορά τι ηθαγένειε στην Σλοβακία. Θα ήθελα επίσης να σα επισημάνω την κατάσταση στη Ρουμανία, όπου ε, δεν τηρούνται οι αρχές ε, του νόμου για την παιδεία σε ό,τι αφορά τις μειονότητες ε, σε πανεπιστήμια και σχολεία. Θα πρέπει να προσέξετε λοιπόν για να μην εστιάσετε σε μία μόνο κυβέρνηση. Ευχαριστώ Σουντία Δημέρα. Δεν είναι παρόν. Και αυτό σημαίνει ότι επόμενος, η επόμενη είναι η κυρία Μπασέσκου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σας επιστήσω την προσοχή σε ένα τραγικό συμβάν, το οποίο πέρασε παρατήρητο φαίνεται στις Βρυξέλλες. Την 1η Ιανουαρίου έλαβε χώρα στην υπερπνησερία ο Μολδαβός, ένας Μολδαβός πολίτης, 18 ετών, σκοτώθηκε σε ένα σημείο ελέγχου από Ρώσο στρατιώτη των ερευνητικών δυνάμεων. Το περιστατικό αυτό κλειδώνει σε όλη την κοινωνία και δημιούργησε σημαντική αβεβαιότητα σε όλη την κοινωνία και αυτό μας υπενθυμίζει ότι στα πρόθυρα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε μία παγωμένη σύραξη και η αποτυχία επίλυση της ε, σύγκρουσης αυτής καθυστερεί την προσέγγιση της Μολδαβίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επίλυση της σύγκρουσης στην Υπερνηστερία προαπαιτεί να δοθεί μια διεθνή εντολή ειρνευτική αποστολή και θέλουμε πιο έντονη ε, δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, κυρία Τσικάου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε η διακυβερνητική συμφωνία που υπεγράφει από 25 κρατημέλη ε, στις 30 Ιανουαρίου αποτελεί μια δέσμευση για πιο έντονη δημοσιονομική πειθαρχία. Δυστυχώς δεν υπάρχει σχετική συμφωνία εξίσου αυστηρή σε ό,τι αφορά την απασχόληση των νέων και για την ενίσχυση την παροχή κινήτρων για την οικονομία. Ο αριθμός των ε, οικογενειών στη Ρουμανία που είναι πλέον στα πρόθυρα της φτώχειας έχει αυξηθεί η κυβέρνηση έχει περάσει νόμους για την παιδεία χωρίς να πάρει την έγκριση του Κοινοβουλίου. Και οι Ρουμάνοι πολίτες αποφάσισαν λοιπόν να εκφράσουν την ανησυχία τους και διοργανώθηκαν ε, διαδηλώσεις αυτό είναι σύνηθε πλέον τις τελευταίες τρεις εβδομάδες. Τα να είμαστε σε θέση να εμπιστευόμαστε την πολιτική. Όπως ε, όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, οι Ρουμάνοι πολίτε δεν περιμένουν, δεν προσδοκούν την λιτότητα. Θέλουν σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν από δύο χρόνια η Ολομέλεια με συντριπτική πλειοψηφία ενέκρινε ε, ένα ψήφισμα για τη... τα ορυχεία. Ωστόσο, επικεντρωθήκαμε και επικαλεστήκαμε τότε τις εθνικές αρμοδιότητες και η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει και να απαγορεύσει αυτή την τεχνολογία σε ό,τι αφορά τις εξορίξεις. Τα σε ό,τι αφορά το κιάνιο ότι πριν, στις 30 Ιανουαρίου του 2000 ε, έλαβε η χώρα μια καταστροφή. Θα παρακαλέσω τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, εξ του Κοινοβουλίου, να πει ένα καλό λόγο για μας στην Κομισιόν και στη Ρουμανία, προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή το ψήφισμα αυτό. Γιατί σε περίπτωση καταστροφής θα ήταν τεράστια η καταστροφή, μέγεθος ε, ατομικής βόμβας. Και αυτό θα έβλαπτε και την Ουγγαρία και τη Ρουμανία. Ευχαριστώ. Αυτή τη στιγμή στο Βουκουρέστι η θερμοκρασία είναι 20 βαθμοί κάτω από το 0 και οι πολίτες συνεχίζουν να διαμαρτύρονται τις τελευταίες εβδομάδες. Ε, παρόμοια κατάσταση έχουμε και σε άλλες πόλεις της Ρουμανίας. Οι άνθρωποι αυτοί βγαίνουν παρά το πολύ ψύχο στους δρόμους γιατί έχουν βαρεθεί την ταπείνωση και το, να τους κοροϊδεύουν οι, οι πολιτικοί. Εξανίστανται κατά της περιφρόνησης αυτής που δείχνουν οι πολιτικοί η απόγνωση του οδηγεί στην συνέχιση της διαμαρτυρίας. Πάνω από το 90% του λαού θέλει ε, να πέσει η κυβέρνηση, αλλά η κυβέρνηση συνεχίζει να τροποποιεί τον εκλογικό νόμο και να παρατείνει τη θητεία της ε, καταπατώντας τις δημοκρατικές αρχές και αξίες. Και την επιθυμία του κόσμου θέλει το, το κράτος να επιστρέψει στα χέρια του λαού. Η κυρία Ζάμπορσκα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ανακοινώσω στο Κοινοβουλίο ότι πριν από κάποιες ε, ε ημέρες απεβίωσε η Βαρόνι Ντεφός που ήταν Ολλανδέζα και ήταν πρόεδρος της Διεθνούς Κινήματος χάρη στον οποίο δημιουργήθηκε το Ινστιτούτο για την Διεθνή Έρευνα για την καταπολέμηση της φτώχειας. Η κυρία Ντεφός κατάφερε να οικοδομήσει σταθερές σχέσεις με τον ΟΗΕ και με τον σχετικό εισηγητή για την καταπολέμηση της φτώχειας μετά την πρώτη της εκλογή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκίνησε μια σχετική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να θυμόμαστε ότι η ακραία φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλο τον κόσμο αποτελεί παραβίαση των θεμελιδών δικαιωμάτων. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η χθεσινή συζήτηση που οργανώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τα προβλήματα δημοκρατίας από την κυβέρνηση Μπασέσκου προκάλεσε το ενδιαφέρον των Ρουμάνων και πολλών άλλων συναδέλφων από άλλες χώρες. Το ότι αυτή η συνάντηση οργανώθηκε από τους σοσιαλδημοκράτες και τους φιλελευθέρους αντιπροσωπεύτηκε και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα από πολλούς βουλευτές που αντιπροσωπεύουν και το κυβερνών κόμμα. Η προσπάθεια την οποία έκαναν ήταν να παρεμποδίσουν την εξέλιξη της συζήτησης και να προσπαθήσουν να απαγορεύσουν ουσιαστικά την συνάντηση επιμένοντας σε δευτερεύοντα θέματα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με το υποσυζήτηση θέμα. Για μια ακόμη φορά όμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέδειξε ότι είναι ένα όργανο που δεν ανέχεται τέτοιου είδους συμπεριφορές και οι ε, συμμετέχοντες καταδίκασαν την προσπάθεια των μελών του ΕΛΚ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν όλους τους βουλευτές που πήραν μέρος στη συνάντηση αυτή και θα ήθελα να σας πω όλους ότι οι Ρωμάνοι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους. Ευχαριστώ. Κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η ασφάλεια στη θάλασσα, αυτό είναι το θέμα μου. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Εδώ και δύο εβδομάδες βυθίστηκε ένα αλλιευτικό τη στιγμή που έμπαινε στο λιμάνι με θύματα. Ζη... Εκφράζω τη λύπη μου προς τις Ιρλανδικές και Αιγυπτιακές οικογένειες την ίδια εποχή είχαμε και το πρόβλημα με το μεγάλο κρουαζιερόπλιο στην Ιταλία. Και ίσως αυτό που ονομάζω εγώ ε, τα πλοία του θεάματος να είναι υπεύθυνα για αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι ακολουθούνται πρακτικές οι οποίες είναι αντίθετες με την ασφάλεια των σκαφών και των επιβατών τους. Ε, τίθεται το θέμα του μεγέθους, του καλύτερου μεγέθους. Πριν λίγα χρόνια είχαμε χίλιους επιβάτες, τώρα έχουμε πέντε χιλιάδες. Τελευταίος ο μιλητής, Ευχαριστώ. Σίγουρα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημαντικό νομοθετικό κείμενο είναι η άκτα. Σε μένα μιλάτε κύριε Πρόεδρε. Επαναλαμβάνω, ε, σημαντική αποφασιστική φάση της ομοθετικής διαδικασίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περνάμε για το θέμα το άκτα, το ε, Anti-Counterfeiting Act. Ε, ήμουν από τα πρώτα θύματα της πειρατείας στο ίντερνετ όταν το ντοκιμαντέρ που είχα γυρίσει ε, αντιγράφηκε παράνομα στο ίντερνετ με χιλιάδες αντίγραφα ε, στη δεκαετία του 90. Παρ' όλα αυτά, παρόλο που ήμουν και εγώ προσωπικά θύμα της πειρατείας, είμαι κατά του άκτα, εξαιτίας της αδιαφάνειας των διατάξεων του, εξαιτίας της τεράστιας απειλής ε, που περιλαμβάνει για το ίντερνετ. Γι' αυτό και σε 80 πολωνικές πόλεις, ε, χιλιάδες νέοι κατέβηκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν κατά τις συνθήκες άκτα. Και ε, μάλιστα ε, σε, ένα, μία, σε μία μικρή ιστοσελίδα, μία μικρή ιστοσελίδα διαγράφηκε από το ίντερνετ ε, επειδή ασκούσε κριτική στην κυβέρνηση. Και νομίζω ότι το άκτα δεν θα προστατεύσει την ελευθερία του ίντερνετ. Το αντίθετο, προτιμούμε το ελεύθερο ίντερνετ και είμαστε κατά του άκτα. Κάτω το άκτα ναι στο ελεύθερο ίντερνετ. Το πρόβλημα είναι ότι δεν καθόσαστε στη σωστή θέση και δεν είχα δεν, είχα καταγραφεί, δεν είχατε καταγραφεί. Αλλά πρώτη φορά ήταν η παρθενική μου προεδρία στην, ε, στην Ολομέλη, γι' αυτό και σας έδωσα το λόγο. Έχετε το λόγο και ε, κύριε Σαλαβράκο. Ε, κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι οι έννοιες και λέξεις δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα είναι έννοιες πολύ ταλαιπωρημένες. Με την ίδια ευκολία που τις εξυμνούμε τις παραβιάζουμε. Οι εκπρόσωποι της Τρόικας στην Ελλάδα απαιτούν για τη σύναψη νέου δανείου προς τη χώρα λήψη εξοδοτικών μέτρων κατά της ελληνικής κοινωνίας. Μεταξύ άλλων ζητούν απόλυση 150.000 δημοσίων υπαλλήλων και μείωση μισθών και συντάξεων στον ιδιωτικό τομέα με κατάργηση του κατώτατου μισθού και των συλλογικών συμβάσεων οι απαιτήσει αυτές είναι αντίθετες προς το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των καταστατικών συνθήκων και καθιερώνουν το δικαίωμα στην εργασία και την προστασία της που αποτελούν βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. υπάρχει κύριε πρόεδρε κίνδυνο διάλυσης του κοινωνικού ιστού και αποσταθεροποίησης στην ελλάδα όσον αφορά την πρόταση τοποθέτηση τοποτηρητή στην ελληνική κυβέρνηση σα βεβαιώνω ότι και ανεφάρμοστη είναι αλλά κυρίω είναι προκλητική για του έλληνε. η κρίση θα περάσει κύριε πρόεδρε. όταν περάσει να μπορούμε ο ένα να κοιτάζει τον άλλον. ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστώ για τι ομιλίε σα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Επίτροπο που έμεινε μέχρι τέλος τη συζήτηση. Ε, ευχαριστώ και τους συνεργάτες μας ε, και τους διερμηνείς